διάταξη πρόγραμμα εργασία τη Επιτροπή για το 2016, δήλωση τη Επιτροπή. Θα ήθελα να πω ότι δεν θα έχουμε διαδικασία catch the όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα, ούτε τη διαδικασία τη γαλάζια κάρτα. Λοιπόν, κυρίε και κύριοι, αξιότιμα μέλη, επόμενο ομιλητή είναι ο Αντιπρόεδρο Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο κ. Φραν Τίμερμαντ. Το πρόγραμμά μας το φετινό είναι ότι δεν έχουμε χρόνο για συνηθισμένες εργασίες και οποιοδήποτε, αυτός είναι ο τίτλος μας, οποιοδήποτε εδώ ή στην Ευρώπη που έχει παρακολουθήσει την πρωινή συζήτηση θα συμφωνεί μαζί μου ότι δεν είναι χρόνος για συνηθισμένες διαδικασίες και εργασίες. Γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα κάνει ρεαλιστικές, τολμηρές, εστιασμένες προτάσεις για να ξεπεράσουμε τις κοινέ μας προκλήσεις και να βγούμε δυνατότεροι στο πνεύμα της ευρωπαϊκής ευθύνης και αλληλεγγύης. Οι δέκα προτεραιότητες του Πρόεδρου Γιούνκερ είναι δήλωση αποστολής μας και είναι και η βάση μας. Έτσι διοριστήκαμε από εσά, με βάση αυτούς τους στόχους. Είναι σωστή στόχη. στόχοι. Πέρσι είπαμε ότι θα κάνουμε διαφορετικά πράγματα και ότι θα κάνουμε τα πράγματα διαφορετικά. Επικεντρωνόμεθα επί των μεγάλων στόχων. Καθορίζουμε όραμα και συγκεκριμένα μέτρα που είναι αναγκαία σε διάφορους ε, τομείς επενδυτικό σχέδιο, ψηφιακή ενιαία αγορά, ενεργειακή ένωση, ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την ασφάλεια, ευρωπαϊκό θεματολόγιο για τη μετανάστευση, κεφαλουχικέ αγορέ, ένωση αυτών, σχέδιο δράση για δίκαιη φορολόγηση ε, των εταιριών. Θέλουμε καλύτερη νομισματική και οικονομική ένωση, πιο ισχυρή και αύριο θα παρουσιάσουμε και τη στρατηγική για την ενιαία αγορά. Φέτος ακόμα θα ολοκληρώσουμε την εικόνα με τα σχέδιά μας για βιώσιμη κυκλική οικονομία, κινητικότητα κατοργατικού δυναμικού και καλύτερη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων. Λοιπόν, το πρόγραμμα εργασία που εθέτησε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι 23 βασικές πρωτοβουλίε εστιάζονται επί υλοποιήσεω των αλόγων στρατηγικών, αντιπροσωπεύει ουσιαστικό ε, νομοθετικό ε, θεματολόγιο και θα υπάρχει πολλή δουλειά για το Κοινοβούλιο όλοι θα λάβατε ένα αντίγραφο ζεστό ζεστό από το τυποτήριο από την πρέσα. Ε, δεν είμαι σίγουρος το διαβάσατε όλοι το πρόγραμμα και γι' αυτό θέλω να αναφερθώ ε, σε πέντε σημαντικά θέματα που θα ήθελα να τονίσω όλους ιδιαίτερος. Λοιπόν το πρώτο ε, θα συνεχίσουμε να θέτουμε προτεραιότητα ε, όσον αφορά τη μετανάστευση και τους πρόσφυγες. Το Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο για τη Μετανάστευση ε, δίνει μια πλήρη απάντηση. Άμεσες δράσεις έχουν αναλυφθεί και είμαι ευγνώμων, πολύ ευγνώμων προς το Κοινοβούλιο και τον Πρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου για την ταχύτητα με την οποία δράσατε και για το ότι ηγηθήκατε ε, συνεχώ ε, όσον αφορά την αντιμετώπιση του θέματο. Προτείνουμε νέα μέτρα για την βελτίωση διαχείριση τη μετανάστευση, ούτω ώστε να αλλάξει και το σύστημα του Δουβλίνου για το άσυλο, να ανανεωθεί και να έχουμε και μια νέα προσέγγιση για την νόμιμη μετανάστευση. Αυτό θα συμπληρώνει τι προτάσει για ενισχυμένη διαχείριση των συνόρων που θα υποβληθούν μέχρι τέλο του έτου μαζί και με μια Ευρωπαϊκή Αρχή για την Προστασία των Συνόρων και Ακτοφυλακή. Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε το θέμα της ανάπτυξης των επενδύσεων και των θέσεων απασχόλησης. Το επενδυτικό ταμείο είναι λειτουργικό, χάρη και πάλι στις προσπάθειες του Ευρωκοινοβουλίου και στην ταχύτητα με την οποία κινήθηκε και δίνει ποιοτικέ επενδύσεις για να τονώσουν περαιτέρω την ευρωπαϊκή οικονομία και την έρευνα. Εστιαζόμεθα επιβελτιώσεως του επενδυτικού περιβάλλοντος και εμβανθύνσεως της ενιαίας αγοράς, ούτω ώστε να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα, λιγότερους φράγμους και σωστό περιβάλλον για καινοτομία, κυρίως μεταξύ μικρομεσών επιχειρήσεων και νεοφιών επιχειρήσεων. Θα κάνουμε συγκεκριμένες προτάσεις, ούτω ώστε να εφαρμοστεί η ενιαία ψηφιακή αγορά και σχετική στρατηγική θα παρουσιάσουμε και τομεακές στρατηγικές για το διάστημα και την ε, άμυνα. Τρίτον, ηγείται η Ευρωπαϊκή Ένωση στις συνομιλίες των Παρισίων για το κλίμα και θα ακολουθήσουν τρει σημαντικές δέσμε μέτρων στα πλαίσια της ενεργειακής Ενώσεω θα δώσουμε ένα πακέτο για κυκλική οικονομία για να μεγιστοποιήσουμε την αποδοτικότητα των πόρων ε, σε όλη την αλυσίδα την οικονομική και θα καθορίσουμε νέες προσεγγίσεις για να εξασφαλίζουμε το ότι οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά θα είναι βιώσιμη η Ευρώπη λαμβάνοντας υπόψη τους, στόχους, τους αναθεωρημένους στόχους για το 2020 και τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ. Τέταρτον, θέλουμε το 2016 να είναι ένα έτος πραγματικής κοινωνικής ε, προόδου. Θα παρουσιάσουμε ένα νέο πρόγραμμα για με στόχο να βελτιώσουμε τις δυνατότητες των ανθρώπων να βρουν εργασία, κυρίως στην τομέα των ψηφιακών. Ε, θα καθορίσουμε νομοθετικές και μη νομοθετικές δράσεις για να δώσουμε ε, μια νέα ε, όθηση στην ισορροπία οικογενειακής ζωή και ζωή στον τόπο εργασία και να στηρίξουμε τις γυναίκες. Και οι προτάσει για τη μετακίνηση του εργατικού δυναμικού, για την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού θα βοηθήσει τον κόσμο να μπορεί να μετακινείται ελεύθερα και θα αντιμετωπιστούν οι καταχρήσει όσον αφορά τα επιδόματα και το κοινωνικό dumping. Ελεύθερη και κίνηση δεν θα πρέπει να απειλεί την κοινωνική προστασία. Το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο του 2016 θα εστιάζεται περισσότερο σε οικονομική και φορολογική κατάσταση που επικρατεί στην Ευρωζώνη και στις κοινωνικές και εργατικές ε, επιδόσεις των κρατών μελών και θα αναπτύξουμε έναν πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο που θα εξυγχρονίζει και θα καλύπτει τα κενά όσον αφορά την νομοθεσία επικοινωνική προστασία και θα εντοπίζει κοινωνική βαθμολόγηση που βασίζεται σε βέλτιστε εθνικέ πρακτικέ, ούτω ώστε να έχουμε μια σύγκληση ε, ανωδική, ε, κυρίω στην Ευρωζώνη. Και Πέμπτον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πιέσει για περαιτέρω πρόοδο προ δίκαια αποτελεσματική και φορολόγηση των επιχειρήσεων που θα είναι ε, φιλική προς την οικονομία. Δηλαδή θα πρέπει να καταβάλουν φόρους οι εταιρείε στη χώρα εκείνη που παράγουν κέρδη. Θα παρουσιάσουμε μια σειρά μέτρων για να διευρύνουμε την, ε, να αυξάσουμε τη διαφάνεια του φόρου των επιχειρήσεων και να αποφύγουμε την φόρο αποφυγή και σχέδιο δράσης για πιο αποτελεσματική ε, αποτελεσματικό καθετός, καθεστώς ΦΠΑ που θα αποφύγει τις απάτες. Ήθελα να τονίσω κάποια στοιχεία εδώ, δεν πάω να παρουσιάσω τα πάντα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεχίσει να εφαρμόζει το Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο Ασφαλεία, η καταπολέμηση τη τρομοκρατία και του οργανωμένου εγκλήματο και θα δώσουμε συνέχεια όσον αφορά τη στρατηγική για το εμπόριο και τι επενδύσει. Και την έκθεση για πιο ανθεκτική και ευημερή νομισματική ένωση. Έχουμε όλε αυτέ τι προκλήσει λοιπόν. Άρα είναι σημαντικό να χρησιμοποιήσουμε όλου του πόρου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ο προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω θα πρέπει να έχει στόχο αποτελέσματα και η ενδιάμεση αναθεώρηση του πολιτικού δημοσιονομικού πλαισίου θα εξετάσει πώ να έχουμε καλύτερου στόχου όσον αφορά τη χρηματοδότηση βάσει προτεραιοτήτων. Δηλαδή να εξασφαλίζουμε ότι η χρηματοδότηση εστιάζεται επί προτεραιοτήτων, όπω είναι η κρίση των προσφύγων, και να εστιαζόμεθα περισσότερο στην επίτευξη των αποτελεσμάτων. Οι προκλήσεις και τα προβλήματα όπως είναι η μετανάστευση, η πρόσβαση στην ενέργεια και στους άλλους πόρους και η αλλαγή του κλίματος, όλα αυτά δείχνουν ότι υπάρχει μια ανάγκη για αποτελεσματική εξωτερική διάσταση, ούτως ώστε να πετύχουμε τους στόχους που εφαρμόζουμε και στην εσωτερική πολιτική. Σήμερα περισσότερο ποτέ δεν γίνεται διάκριση μεταξύ εσωτερικών και εξωτερικών προβλημάτων και στόχων. Ήθελα να αναφερθώ στου στόχου τη βιώσιμη ανάπτυξη, που εκεί που δεν μπορεί να γίνει διάκριση μεταξύ εσωτερικού και εξωτερικού. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συμβάλλει σημαντικά στη νέα παγκόσμια στρατηγική και για την στρατηγική της ασφάλειας. Και εδώ ε, πάνε χέρι, με χέρι εσωτερική και εξωτερική διάσταση. Δύο τελικά στοιχεία. Το πρώτο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είπε ότι θα κάνουμε τα πράγματα με διαφορετικό τρόπο. Όλες οι δράσεις που προτείνουμε στηρίζονται στο πρόγραμμά μας για καλύτερη θέση νομοθεσίας. Είμαστε αφοσιωμένοι στην προσπάθειά μας. Όταν θα παρεμβαίνουμε σαν Ευρωπαϊκή Ένωση θα κινούμεθα με τέτοιο τρόπο που θα πετυχαίνει αποτελέσματα και θα κάνει τη θετική διαφορά επιτόπου. Το πρόγραμμα εργασιών όμως συμπεριλαμβάνουμε και τα σχέδιά μα να ανθερήσουμε βασικού τομεί τη υφιστάμενη νομοθεσία, όπω υγεία και ασφάλεια στον τόπο εργασία. Να εξασφαλίσουμε ότι πετυχαίνουν το σκοπό του και συνεχίζουν να έχουν αποτελέσματα όσον αφορά τη φιλόδοξη πολιτική μα και του στόχου προτείνουμε και σειρά αποσύρσεων πρωτοβουλειών που έχουν γίνει απειρχιωμένες ή έχουν αποδυναμωθεί και δεν έχουν πιθανότητες να υιοθετηθούν. Ο κατάλογος είναι αρκετά βραχύτερος από πέρσι που ήταν μια στιγμή διακοπής πολιτικής λαμβάνοντας υπόψη και τη δέσμευση που αναλάβαμε στη Συμφωνία Πλαίσιο που θα κάνουμε αυτές τις αποσύρσεις και ανακλήσεις από τη στιγμή που θα ακούσουμε τις δικές σας απόψεις. Δεύτερο σημείο. Το πρόγραμμα εργασίας δεν μπορεί να πετύχει αποτελέσματα χωρίς επαρχή ε, συμμετοχή των συνομοθετών να το στερνιστούν το πρόγραμμα δηλαδή. Και εδώ ε, χρειάζονται τρει για να χορέψουν και είναι περίεργο αυτό. Το πρόγραμμα εργασιών ε, καλύπτεται από το δικαίωμα πρωτοβουλία Ευρωπαϊκή Επιτροπή και φέρουμε την ευθύνη. Δεχόμαστε την ευθύνη για τι προτάσει. Για να είναι ισχυρή η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να μπορεί να αποδείξει ότι όλοι οι θεσμοί μα είναι έτοιμοι να ετοιμάσουν το αιματολόγιο τη Ευρώπη μαζί και να συνεργάζονται γρήγορα και να θέλουν να πετύχουν του στόχου μα. Προετοιμάζοντα το πρόγραμμα εργασιών, λάβαμε υπόψη τι απόψει που εκφράσατε εδώ και το ψήφισμά σα και νομίζω ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλος βαθμός συγκλήσεως. Όλοι θα συμφωνούν, θαρώ, ότι οι κοινέ μέθοδοι εργασίας για τον φετινό διάλογο έχουν βελτιωθεί κατά πολύ. Έχουμε ε, ε, έχουμε τις συζητήσεις CCC και το νέο, ε, το νέο σύστημα που ακολουθούμε και ευχαριστούμε για όλες τις προτάσεις των Επιτροπών σας και των Πρόεδρων των Επιτροπών καθώς και των ομάδων και των ηγετών των ομάδων. Ευχαριστώ όλους τους ηγέτες των ομάδων γιατί ηγήθηκαν σε αυτό το τομέα. Ευχαριστώ τον Πρόεδρο Σούλτς που πήρε πολύ σοβαρά το θέμα και μας βοήθησε να οργανώσουμε καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο συνεργαζόμαστε και εργαζόμαστε και ευχαριστώ και τον πρόεδρο Μπούζεκ που ανέλαβε την ευθύνη να κάνει το ίδιο με το σύστημα CCC. Ελπίζω λοιπόν όλα αυτά να μας βοηθήσουν να καταλήξουμε σε κοινή κανανόηση των προτάσεων των τωρινών και των μελλοντικών και ελπίζουμε οι συνομοθέτες να ε, κινηθούν γρήγορα. Προσβλέπω σε συνεργασία μαζί σας και το 2016 και χαίρομαι που μπορέσαμε να βελτιώσουμε τις μεθόδους εργασίας προς ικανοποίηση ελπίζω ε, και των δύο θεσμικών μας οργάνων και σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε μας Για το ΕΛΚ. έχει τον λόγο κύριο Σάγερ παρακαλώ. Ε. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε. Μετά από μεγάλο διάστημα διαπραγματεύσεων το Σεπτέμβριο συμφωνήσαμε μεταξύ διαφορετικών εταίρων σε αυτό το σώμα και ήταν ευρύτερα θεμέλια αυτά για το έργο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ανακοινώθηκε και αυτό σε σχέση με την Επιτροπή. Και λόγω της συμφωνίας δεν υπάρχει κάποια μεγάλη ένταση. Ε, αν υπήρχε καταψήφιση δεν θα υπήρχε συμφωνία και τότε θα υπήρχε πολύ μεγαλύτερη αντίδραση. Είναι όμως πάρα πολύ σημαντικό το Ευρωκοινοβουλίο και η Επιτροπή να συνεργαστούν από κοινού, διότι η Ευρωβουλή ε, όταν εξελέγει το μήνυμα για το πώς εργάζονται τα θεσμικά όργανα θα πρέπει να αλλάξει σημαντικά. Πρέπει να είναι πολύ πιο αποτελεσματικά τα θεσμικά όργανα. Ένας μικρός κατάλογος μπορεί να αναφερθεί από πλευράς του ΕΛΚΑ για τους τομείς όπου μπορεί να υποστηριχθούν οι κατευθύνσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής από πλευράς μας. Μεθοδολογικά ιδιαίτερα. Καλοχαιρετίζουμε την συμπίκνωση των 10 προτεραιοτήτων του συστήματος του προγράμματος Juncker από πλευράς μας. Αναλογικά επίσης ε, το κλειδί πρέπει να ευθυγραμμίζεται με την επικουρικότητα και την αναλογικότητα. Και <clears throat> είδαμε ευρύτατα και μεγάλα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά το παρελθόν που δεν υλοποιήθηκαν. Η υλοποίηση λοιπόν, η αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας, η εξέταση και εκτίμηση επιπτώσεων, η παρακολούθηση καθ' όλη τη διάρκεια ε, των ε, προγραμμάτων και των ε, πρωτοβουλειών είναι κάτι πολύ σημαντικό. Και μεθοδολογικά πάλι ζητούμε να ευθυγραμμίσει την νομοθεσία σε σχέση με τις κατεντολήν πράξεις και κατεξουσιοδότηση πράξεις η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το ε, θέμα αυτό είναι πολύ μεγαλύτερο ωστόσο και είναι κάτι το οποίο εξετάζουμε και μετά από πολλά χρόνια μετά την έγκριση της συνθήκης Λισαβόνας θα πρέπει να επικεντρωθεί στην ε, υλοποίηση της ε, ενισχύ νομοθεσίας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κάνουμε λόγο για την κοινή αγροτική πολιτική για παράδειγμα ή την κοινή πολιτική συνοχής. Υπάρχουν δύο προτεραιότητες σε αυτόν τον τομέα που θεωρεί πάρα πολύ σημαντικές ως υποθέσεις το ΕΛΚΑ. Η κινητικότητα και η ελαστικότητα της αγοράς εργασίας πρέπει να βελτιωθούν, καθώς και η απασχόληση των νέων. Και πρέπει να βελτιωθούμε ώστε να έχουμε καλύτερη, καλύτερα αποτελέσματα και όσον αφορά και την καινοτομία. Πρέπει να ολοκληρωθεί και η ενιαία αγορά, πράγμα το οποίο είναι προτεραιότητα και στον ενεργειακό τομέα και στον ψηφιακό τομέα. Η ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων είναι πολύ σημαντική υπόθεση υπόθεση, ιδιαίτερα των μικρομεσαίων ε, επιχειρήσεων, είναι μεγάλη προτεραιότητα για να διασφαλιστούν και να διασωθούν θέσει απασχόληση ε, στην Ευρώπη. Ωστόσο, η κατεπίγουσα αντιμετώπιση τη κρίση ε, των προσφύγων είναι κύρια πρόκληση. Πρέπει να υπάρχουν ασφαλή εξωτερικά σύνορα, θεωρεί το ΕΛΚ, να αντιμετωπιστούν οι κίνδυνοι. Πρέπει να διασφαλιστεί η ασφάλεια των πολιτών μα. Αυτή πρέπει να είναι και είναι η κύρια προτεραιότητά μα. Και το Κοινοβούλιο έχει ήδη καταδείξει την προθυμία του να συνεργαστεί και να δράσει άμεσα και ταχύτατα επ' αυτών. Καλωσορίζουμε λοιπόν τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, για το πρόγραμμα εργασίας, εργασιών του 2016. Ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε πολύ λέει ο Πρόεδρος κύριε Σάιερ. Για την Σοσιαλδημοκρατική Ομάδα Ροντρίγε παρακαλώ. Yes, ε, Mr. Vice President. Μάλιστα κύριε Αντιπρόεδρε. Βέβαια και δεν είναι ρουτίνα η, αυτό το πρόγραμμα. Τα όσα λέτε είναι έγκυρα, αλλά πρέπει κατά τη γνώμη μου να διαρθωθούν με τελείως διαφορετικό τρόπο. Θεωρούμε ότι η βασική κεντρική μας πρόκληση αυτή τη στιγμή είναι η κρίση του η προσφυγική. Να παρεμποδίσουμε την ανθρωπιστική κρίση με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορέσουμε ταυτόχρονα να προστατεύσουμε το χώρο Σέγγεν. Και ξέρουμε ότι αυτό απαιτεί ένα πραγματικό σύστημα ασύλου στην Ευρώπη, ένα πραγματικό ευρωπαϊκό σύνορο και πραγματική ε, μεταναστευτική πολιτική. Οπότε η δική σας επιτροπή θα πρέπει να ε, οικοδομήσει αυτά τα μέσα. Ταυτόχρονα όμως θα πρέπει να μετατρέψουμε την Ευρώπη σε ένα πραγματικό χώρο ευημερία. Και πιστεύουμε πως φέτος θα πρέπει η Κομισιόν να ανανεώσει τη στρατηγική της Ευρώπης 2020 με τρόπο ώστε να μην πρόκειται μόνο για την ενεργειακή μετάβαση αλλά για την ε, οικονομία, την κυκλική, ώστε να διαχειριστούμε καλύτερα τους πόρους μας. Δεν πρόκειται μόνο για έρευνα και ανάπτυξη, αλλά για προσπάθεια εξέβρεσης ε, καινοτόμων λύσεων για να δημιουργηθούν θέσεις απασχόλησης ποιοτικέ. Και ε, μέσω της αναθεώρησης των δημοσιονομικών μέσων μας να μπορέσουμε να αποδώσουμε περισσότερο σε, αυτές, σε αυτή τη στρατηγική. Ταυτόχρονα όμως μας ανησυχεί κάτι που συμβαίνει τώρα στην Ευρώπη. που είναι μια κούρσα προς τα κάτω. Τα κράτη-μέλη ανταγωνίζονται μεταξύ τους, υποβαθμίζοντας τις κοινωνικές προδιαγραφές τους. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να έχουμε έναν ισχυρό πυλώνα για τα κοινωνικά δικαιώματα, ε, για ένα πακέτο κινητικότητας που θα έρθει, αλλά είναι ταυτόχρονα η κατάλληλη στιγμή να, αντιμετωπίσουμε την φοροδιαφυγή με τέτοιο τρόπο, όπου, ώστε οι φόροι να καταβάλλονται εκεί όπου ε, γίνονται τα κέρδη. Θεωρούμε ότι και αυτό είναι μεγάλη προτεραιότητα και Πιστεύουμε ότι αυτή η φιλοδοξία για ολοκλήρωση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης θα πρέπει να καθοδηγείται από ένα κεντρικό στόχο που θα είναι η σύγκληση προς τα πάνω. Κύριε Αντιπρόεδρε, θεωρούμε ότι αν θέλουμε όντως να επιτύχουμε αυτή τη σύγκληση προς τα πάνω θα πρέπει να ολοκληρώσουμε την Τραπεζική Ένωση αλλά και να φτιάξουμε και μια πραγματική δημοσιονομική δυνατότητα εντός Ευρωζώνης. Όλες αυτές οι φιλοδοξίες όμως δεν θα είναι αποτελεσματικές εάν δεν υποστηριχθούν από και πιο φιλόδοξη εξωτερική δράση. Αυτό είπατε. Ναι, συμφωνούμε μαζί σας ότι πρέπει να έχουμε μια παγκόσμια στρατηγική ε, ενημερωμένη, εξυγχρονισμένη και πρώτο ε, ε, το πρώτο έργο της θα είναι να ηγηθεί η Ευρώπη της διάσκεψης του Παρισιού, ε, να ηγηθεί στην επίτευξη των βιώσιμων στόχων, αλλά και να ηγηθεί στην πραγματική εταιρική σχέση με την Αφρική, που είναι η γειτονική μας Ήπειρος. Αυτές είναι οι προσδοκίες μας για τα επόμενα χρόνια. Το Κοινοβούλιο μας θα είναι πολύ δραστήριο στο ψήφισμα και μπορείτε να είστε βέβαιος ότι θα εξακολουθήσουμε, εξακολουθήσουμε να είμαστε δραστήριοι... και θα οθήσουμε προς την κατεύθυνση. Σας ευχαριστούμε κυρία Ζωά Ροντρίγκες. Τώρα για την ECR Ford παρακαλώ. Thank you. Ευχαριστώ. Πρέπει να εστιάσουμε στην πρόθεση της ανταγωνιστικότητας καινοτομία και του εμπορίου σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, στον νέο ώρα και την ψηφιακή αυτή εποχή και θα πολλά στο πρόγραμμα εργασιών ε, με βρίσκουν σύμφωνοι είπα ότι κάθε πρωτοβουλία τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω πρέπει να εστιάζεται επί του στόχου. Θα διευκολύνει, θα δυσχεραίνει τι επιχειρήσει των ανθούν. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει περικόψει την τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω, εξασφαλίζει ότι οι ισχύοντε νόμοι θα λειτουργούν και υποσχεθήκατε να μειώσετε τη γραφειοκρατία και αφαιρέσατε 70 προτάσει. Ευχαριστώ, Επίτροπε, που εισακούσατε τα όσα είπε το ECR. Όμω το ψήφισμα του Κοινοβουλίου για το πρόγραμμα εργασία ζήτησε μια βαθύτερη πολιτική ένωση και ευρωπαϊκά πρότυπα για την ευημερία, την προστασία τη υγεία και την παιδεία και διαφωνώ. Αυτά είναι θέματα που τα διευθετούν καλύτερα οι εθνικέ κυβέρνησει και ξέρω ότι πολλοί συνάδελφοι στο Κοινοβούλιο είχαν την ίδια άποψη. Η ενιαία αγορά έχει σαν στόχο να βοηθήσει τη δημιουργία οικονομικών δυνατοτήτων που οδηγεί σε ανάπτυξη και θέσει εργασία. Είπατε ότι τώρα δεν είναι χρόνο για συνηθισμένη προσέγγιση στα θέματα. Ας μην ξεγελαστούμε από την αριστερά και κάνουμε προτάσεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μια κατάσταση στην οποία η Ευρώπη δεν μπορεί να κινηθεί σωστά όσον αφορά τις επιχειρήσεις. Ευχαριστούμε για τους φιλελευθέρους η κυρία Ιντφέλτ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Νομίζω δεν είναι η κανονική δουλειά που θα συνεχίζεται ως συνήθως, διότι κατάφερε ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κάτι επαναστατικό, να επικεντρώνεται σε ουσιώδη θέματα το πρόγραμμα της εργασιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σας συγχαίρω γι' αυτό. Δεν είχα πραγματικά τον χρόνο να διαβάσω σε λεπτομέρειες ε, το πρόγραμμα αλλά ρίχνοντας μια ματιά σημειώνω πολύ θετικά πράγματα που θα έχετε για αυτά την υποστήριξη της ομάδας μας και για το κεφάλαιο της μετανάστευσης και του ασύλου και τις προτάσεις ε, για μια ακτοφυλακή που θα ε, μπορέσουν να αναζωογονήσουν ε, και την κιανή, την μπλε κάρτα και την ισορροπημένη προσέγγιση ώστε να μπορεί να δρά η Ευρώπη και για τις επίσης ε, και την, πρόταση για την εξωτερική εκπροσώπηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και υπάρχουν πολλά περισσότερα θέματα τα οποία θα υποστηριχθούν από πλευράς μας οπωσδήποτε. Κάποια πράγματα όμως απουσιάζουν νομίζουμε και έχουμε και κάποια ερωτηματικά σχετικά. Ένα από τα πράγματα που θα θέλαμε να ενταχθούν και ζητήθηκε από το Ευρωκοινοβούλιο όταν γινόταν λόγος για την, το κεφάλαιο ασφάλειας είναι το ότι κατεπηγόντως χρειαζόμαστε εδώ και χρόνια τώρα μία σε βάθος εξειδικευμένη αξιολόγηση των μέτρων που υιοθετούνται και την αποτελεσματικότητα αυτών. Πόσο αποτελεσματικά είναι. Είναι πράγματι μέρος της καλύτερης νομοθεσίας και καλύτερης νομοθετικής δράσης. Κάπως για παράδειγμα παράδειγμα η αποτροχοπέδηση της εγκάρσιας οδηγίας κατά των διακρίσεων και υπέρ των ε, γονεϊκών θεμάτων. Είναι θέματα για τα οποία είναι υπέρ το Κοινοβούλιο και έχουμε την τιμή να εκπονήσουμε και να προτείνουμε ένα μηχανισμό για τα θεμελιώδη δικαιώματα, την ε, ε, δημοκρατική διακυβέρνηση και τέλος ε, για την ψηφιακή ημερήσια διάταξη, για το ψηφιακό θεματολόγιο. Καλωσορίζουμε το έργο σας. Αλλά πώς να ερμηνεύσουμε τα όσα είπε ο κύριος Έτιγκερ, αντί να υπάρξει δημιουργία ενός παγκόσμια ανοιχτού διαδικτύου, να μπορέσουμε να επικεντρωθούμε σε σχέση με ένα ευρωπαϊκό ε, σύστημα νεφοϋπολογιστών και δεν γνωρίζω αν εσείς συμφωνείτε με αυτές τις προτάσεις ή όχι. Δεν πρόκειται εδώ μόνο για την έκβαση της πολιτικής συζήτησης αλλά για την ίδια τη διαργασία και διαδικασία. Πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πολλά περισσότερα θα μπορούσε να πράξει. Παράδειγμα, διαφάνεια. Θα μπορούσαμε πολλά περισσότερα να κάνουμε για να γίνουμε προπομπή, πρωτοπόροι, να μπορέσουμε να βρεθούμε στην πρώτη γραμμή ε, των των και όχι να γίνονται όλα αυτά και κλεισμένων των θυρών, εγκρυπτό και παραβίστο. Πρέπει επίσης να εξετάσουμε την ποιότητα του νομοθετικού έργου και επίσης να εξετάσουμε και τους ίδιους τους εαυτούς μας με πιο κριτικό πνεύμα. Βαρέθηκα και κουράστηκα σε σχέση με τα πράγματα όσα έχουν με νομοθετικό έργο το οποίο δεν βαίνει καλός και, ε, και έχει σαθρά θεμέλια και θα καταλήξει στο τέλος τέλος με προσφυγές στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Μεγαλύτερη έμφαση να δώσουμε στις διεργασίες. Η τελική έκβαση είναι φυσικά στο τέλος τέλος πολιτική επιλογή, θέμα πολιτικής επιλογής και κριτηρίων. Αλλά το πώς θα αντιμετωπίζουμε σε διεργασίες και διαδικασίες αυτά τα πράγματα είναι κάτι του οποίου πρέπει να συμφωνήσουμε όλοι. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για την Ενωτική Αριστερά. Η κυρία Μίχελς τώρα παρακαλώ. Η ε, Κυρία Μίχελς, κύριε Πρόεδρε, ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Γιούγκερ σήμερα το πρωί στο Κοινοβούλιο μίλησε και χρησιμοποίησε πραγματικά λόγια που μας συγκίνησαν για την πολιτική ε, για τους πρόσφυγες. Όμως ε, ποιες είναι οι θαραλές επιπτώσεις ε, το ότι κρατάμε ακόμα μια παροχημένη ιδεολογία ανταγωνισμού για τον, ε, τις ιδιωτικοποιήσεις και για το πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων του κ. Γιούγκερ όχι, δεν μπορούν να γίνουν αυτά. Ανισότητες κοινωνικές είναι τα θεμέλια της απόρριψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πολλές φορές και για ρατσισμό. Καλά θεμέλια για την πολιτική ανάπτυξης και απασχόλησης, για την κοινωνική και πολιτισμική ολοκλήρωση και ένταξη και την προστασία των προσωπικών δεδομένων και των καταναλωτών. Στο τέλος τέλος παραμένουν στις προτάσεις σας λεπτομέρειες και προγράμματα διορθωτικά επιδιορθώσεων δεν χρησιμοποιούνται, δεν έχουν ε, ε, κανένα όφελος και οι καλύτερες ιδέες όταν οι αρχές της ελευθερίας, ισότητας και αλληλεγγύης παραμένουν ωραία κενά λόγια σε δεκάρικους λόγους ε, και σε κατηχητικές τέτοιες παρεμβάσεις. Χάσατε δυστυχώς την ευκαιρία κύριοι της Επιτροπής, δεν την εκμεταλλευτήκατε. Πρόεδρος. Τον λόγο θα λάβει τώρα για την ομάδα των Πρασίνων ο κύριος Λάμπερτς. Κύριε, Πρόεδρε, κύριε Αντιπρόεδρε, καλώς ορίσατε. Παρατήρησα στη διάρκεια του 2014 και κυρίως του 2015 ότι η Επιτροπή κυρίως απέναντι στην πρόκληση που παρουσιάζει η ροή των μεταναστών προς την Ευρώπη ενεργεί με ε, φιλοδοξία ε, και γρήγορα. Πάντως, ε, ορισμένοι παραμένουν ανικανοποίητοι, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν κάνετε αυτό που έπρεπε. Θα ήθελα όμως πραγματικά να κάνετε το ίδιο για τα ζητήματα που απασχολούν τους Ευρωπαίους, γιατί άκουσα πολύ καλά τον κατάλογο προτάσεων που θα μας υποβάλλετε. Η πυκνότητά τους ε, αντιστοιχεί στην ε, πυκνότητα των μελών μέσα σε αυτή την αίθουσα. Για το 2014 κάνατε την εξαρτία και όλοι αισθανθήκατε ότι το θέμα αυτό είναι κρίσιμο για τους Ευρωπαίους. Η Κομισιόν ε, το 2014 ανέλαβε καθήκοντα ε, το 2014 και μέχρι στιγμής για αυτό το θέμα δεν έχει γίνει τίποτα. Αλλά δεν είναι αλήθεια ότι δεν έχει γίνει τίποτα ε, γιατί η αναχώρα συστάσεις στο πλαίσιο των εξαμήνων εξακολουθούν να προχωρούν προς την ίδια κατεύθυνση. Δηλαδή επιδεινώνουν το κοινωνικό ντάμπινγκ ανάμεσα στα κράτη-μέλη μέσω των μεγαλύτερων, ε, της μεγαλύτερης ευελιξίας που συστήνουν κτλ. Ε, τώρα, φορολογική ω ανταγωνισμό. Πριν από ένα χρόνο είχαμε το σκάνδαλο LuxLeaks. Έκτοτε ένα μικρό, ε, ένα μικρό μέτρο, ανταλλαγή πληροφοριών για τα tax ruling. Ε, μέτρο το οποίο αποδυναμώθηκε από το Συμβούλιο που λάμπει δια τις απουσίας του εδώ. Και μας λέτε ναι, ναι, αύριο μανιάνα η λύση. Εκεί δεν φαίνεται να έχετε μεγάλες φιλοδοξίες λοιπόν για το κοινωνικό, φορολογικό και περιβαλλοντικό dumping, αυτά που θέλετε με το TTIP και με την καλύτερη νομοθεσία προχωρούν προς την αντίθετη κατεύθυνση από αυτή που θα έπρεπε για την Ευρωζώνη. Ξέρετε ότι έχει μπλοκαριστεί στο Συμβούλιο. Μα τι περιμένετε για να υποβάλλετε προτάσεις που να τοποθετήσουν τα κράτη-μέλη ενώπιον των ευθυνών τους. Ε, ε, ε, αυτόματος αθεροποιητής προϋπολογισμός της Ευρωζώνης. Ε, εσείς έχετε το δικαίωμα πρωτοβουλία, χρησιμοποιήστε το. Για την υπόθεση του Volkswagen περίμενα πραγματικά να ενεργήσει. Είναι σκάνδαλο για τη δημόσια υγεία, για το περιβάλλον, για το σεβασμό του, του, νόμου. Στρέβλωση της αγοράς, θέματα για τα οποία είναι αρμόδια η Κομισιόν και τι μας λέει η Επίτροπος Βιανκόφσκα Α, κοιτάξτε, α κάνουν τη δουλειά του τα κράτη-μέλη. Εμεί παρατηρούμε, αλλά μην περιμένετε από εμά να αναλάβουμε πρωτοβουλία. Τι συμβαίνει λοιπόν, η αυτοκινητοβιομηχανία είναι ταμπού. Και ξέρουμε ότι στην Γερμανία είναι ε, ε, καλύτερα εδρεωμένη. Παρακαλώ λοιπόν αλλάξτε στάση, αλλάξτε φιλοδοξίες. Πείστε μας σε ένα χρόνο από τώρα ότι πραγματικά καταλάβατε πόσο μεγάλες είναι οι προκλήσεις. Σας ευχαριστούμε. Στη συνέχεια ο κύριος Μπορέλη παρακαλώ. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Σήμερα η Ευρωπαϊκή ε, Επιτροπή ε, έκανε εδώ συνεδρίαση και μας παρουσιάζει το πρόγραμμα για το 2016 και προσπαθεί να μας πείσει ότι δεν πρόκειται για παραδοσιακή διαχείριση. Εγώ θα ήθελα να υπογραμμίσω κάποια οριζόντια και στρατηγικά μέσα που σίγουρα θα απαιτήσουν μη συμβατικά μέτρα. Όποια και αν είναι η πρακτική παρουσίαση του προγράμματος για το 2016 θα πρέπει να δούμε τι έγινε το 2015. Καταρχήν το μάθημα που αποκομίσαμε από την Ελλάδα. Πρέπει να προλάβουμε τις δυναμικές που οδήγησαν ένα έθνος της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ζει σε μια μεγάλη και ε, ε, πολύ μεγάλη φτώχεια. Χρειάζονται μέτρα. Συρία, η δυνατότητα να ενεργήσουμε, η διαδυναμία μάλλον να ενεργήσουμε με συγκεκριμένο και στρατηγικό τρόπο μας έθεσε ενώπιον πολύ σοβαρών προβλημάτων. Το δίδαγμα από τη Volkswagen θα πρέπει οι μεγάλοι όμιλοι να ελέγχονται καλύτερα και να παρακολουθούνται και οι ελεγκτές τους που σε αυτή την περίπτωση ε, ε, έκαναν λάθος, απέτυχαν. Τι θα γινόταν άμα πρόκειται για φαρμακευτικά προϊόντα ή για τρόφιμα. Περιμένουμε συγκεκριμένη πρωτοβουλία από πλευρά σα. Έπειτα, τρία θέματα οικονομικού χαρακτήρα που θα μα συνοδεύουν όλοι το 2016. TTIP, Κίνα και ΕΦΣΥ. Για τις μακροοικονομικές πολιτικές, για τις εμπορικές συμφωνίες μεγάλου εύρους θα πρέπει να υπάρχει μελέτη αντικτύπου μη συμβατική. Πολύ συχνά οι Βρυξέλλες έδειξαν, ε, κράτησαν μειοπική στάση γιατί δεν έκαναν ε, κατάλληλη ανάλυση αντικτύπου. Το ίδιο κάνουν και με το με την ε, Κίνα. Θα πρέπει να υπάρξει μελέτη αντικτύπου για την οικονομία μας. Στην Κομισιόν τώρα θα, η Κομισιόν θα πρέπει να κάνει τη σύνθεση και να δείξει σε ποιες χώρες θα λάμψει ο ήλιος και πού θα υπάρξει, ε, πού ο καιρός θα είναι νεφελώδης. Αν υπήρχε άλλη μια χώρα που, καταλήξει σε μια τέτοια μπόρα, δεν θα είναι σωστό αυτό για την υπόλοιπη Ευρώπη. Έπειτα να θυμίσω κάτι όπου είναι σημαντική η θέση της Ευρώπης. Τα τελευταία στοιχεία της Ευρωστάτ δείχνουν ότι ένας στους τέσσερις Ευρωπαίους ζει σε συνθήκες στόχες. Εμείς θεωρούμε ότι μέτρα όπως το μήνυμο εισόδημα και τα, οι μικροπιστώσεις είναι απαραίτητα μέσα για να δώσουμε το μήνυμα μιας Ευρώπης που βρίσκεται είναι ταυτότητά της, της αλληλεγγύης. Και γι' αυτό θα και θεωρούμε και θέλουμε η Ευρώπη να είναι πιο δυνατή μέσα στο 1916. Καλύτερη νομοθεσία θα πρέπει να βγει από, μάλλον να αντιμετωπίσει μια πρόκληση που σημαίνει τη συμμετοχή των τοπικών αρχών Επίσης να δούμε και ποιες είναι οι, ποιος είναι ο αντίκτυπος των γεωγραφικών ε, ζητημάτων. Δημόσια διαβούλευση λοιπόν για όλα αυτά τα θέματα και σας ευχαριστώ για τον χρόνο που μου δώσατε. Στη συνέχεια ο Σαλβίνη παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Στην έρημο αυτή, η έρημο αυτή τη αίθουσα μα φαίνεται ε, πώ η Σοβιετική Ένωση, η Ευρωπαϊκή Ένωση ζει σε άλλο πλανήτη. Η μετανάστευση είναι μια καταστροφή. Σήμερα το πρωί ο πρόεδρο, ο κύριο Γιούνκερ, μα είπε ότι μετά από μένε συζητήσεων και θριάμβων, το αποτέλεσμα που πέτυχε είναι ότι μόνο εννέα χώρε είναι διαθέσιμες να δεχτούν 700 ε, μετανάστες. Μας λείπουν μερικές εκατοντάδες χιλιάδες και κάποιος θέλει να βάλει την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Τουρκία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όχι, η Τουρκία δεν ήταν ούτε ποτέ θα είναι Ευρώπη και κανείς δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τη μετανάστευση σαν εμπόριο ανταλλαγής και για να αποδυναμώσει τα δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών. Δεν ακούγεται τίποτα λοιπόν σχετικά με του ανέμου του πολέμου που φυσούν. Τι θα κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αυτό το Κοινοβούλιο για να σταματήσει να εξοδετερώσει την, το ISIS που εξοδετερώνει εκατοντάδε χιλιάδε ανθρώπου. Θέλουμε να προθωρήσουμε με τι τελέσει οικονομικέ κυρώσει κατά τη Ρωσία που φέτο μόνο η την Ιταλία οδήγησαν σε ζημιέ 2 δισεκατομμύρων ευρώ για την Ιταλία. Και τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Ουκρανία δεν γίνονται πιο σεβαστά από ότι τα δικαιώματα ε, των ανθρώπων στη Συρία που χρηματοδοτούνται από την Πιστεύω ότι, ότι γίνονται κάποιε θυσίε για την εργασία ε, και στι συντάξει και βρίσκει ευελιξία η Ευρώπη μόνο όταν ανακατεύονται οι μεταναστεύονται για την Κίνα και την οικονομία τη αγορά που κάποιο εδώ θα ήθελε να προωθήσει για να κάνει τι εξαγωγέ και να δημιουργήσει και άλλους ανέργους. Τίποτα για την ε, θεσία την υποχρεωτική των διαφόρων ε, προϊόντων που θα προστάτευε τους κατανοτές και τους παραγωγούς που μόνο την Ιταλία δημιουργούν 60 δισεκατομμύρια ευρώ ζημίας. Να βγάλουμε περισσότερες προστασίες που γίνονται στον αφορά τα άτομα. 80.000 τόνοι ρυζιού έρχονται από το Βιετνάμ χωρίς ελέγχους. 35.000 τόνοι ελαιολάδου από την Ισία χωρίς ελέγχους. Περισσότεροι άνεγοι στην Ευρώπη και περισσότεροι άνθρωποι που ε, καταφθάνουν στην Ευρώπη. Κάτι δεν πάει καλά. Ευτυχώ όταν ψηφίζει ο κόσμο, διαλέγει, επέλεξε στη Βιέννη, στην Πολωνία. Του χρόνου θα γίνει δημοψήφισμα στη Βρετανία και θα διαλέξει. Ελπίζω να γίνει επιλογή και στην Ιταλία και μετά θα είναι προφανέ ότι ε, είναι μια, ένα κλουβί ε, η Ευρώπη αυτή και όσο πιο γρήγορα βγούμε από αυτή, αυτό το κλουβί, τόσο καλύτερα για όλου. Κυρία Μορβάη. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ρωτήσω κάτι τον κύριο Φραντ Τίμερμανς, τον αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Λοιπόν, έχω την εξής ερώτηση για αυτόν. Συμφωνείτε μαζί μου ότι αυτά που συμβαίνουν τώρα εδώ σχετικά με το πρόγραμμα εργασιών του 2016 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αυτή η συζήτηση με άλλα λόγια στο Κοινοβούλιο, όπου έχουμε περίπου 20 ευρωβουλευτές παρόντες. Αυτή η συζήτηση λοιπόν σημαίνει Το ίδιο είναι αντιστοιχή συζήτηση που γίνεται εδώ με μια αντίστοιχη συζήτηση που θα γινόταν σε κοινοβούλιο κράτους μέλους, παίρνοντας αυτό σαν παράδειγμα. Προς εξηγείται το ότι αγαπητός μας ε, ηγέτης ο κύριος Γιούνκερ και η Ευρωπαϊκή του Επιτροπή και, και το Ιωνί κυβερνητικό πρόγραμμα που αφορά πάνω από 500 εκατομμύρια Ευρωπαίους πολίτες απεστάλλει 15 λεπτά μόλις πριν από τη συζήτηση στα ερετά μέλη του Κοινοβουλίου μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Λίγα λεπτά πριν τη συζήτηση απεστάλλει, που, τη συζήτηση που ξεκίνησε στι 3. Πώ εξηγείται αυτή η διαδικασία, τελευταία στιγμή, να στέλνονται αυτά τα έγγραφα στους, στα 500 εκατομμύρια Ευρωπαίου πολίτε. Πώ εξηγείται αυτή η διαδικασία, δεν είναι ταπεινωτική. Και εσά και στον κύριο Σούλτ ε, απευθύνω το ερώτημα. Σαν πρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου, κύριε Σούλτ, δεν θα πρέπει να τοποθετηθείτε από αυτού. Θεωρητικά ήθελα να συζητήσω τη μεταναστευτική πολιτική, που είναι αποκλειστικά είναι μόνο ένα κεφάλαιο αυτού του πρόχειρου προγράμματο. σω κατά τη διάρκεια του διαλύματο για το γεύμα γράψατε πέντε πράγματα γιατί πρέπει να κάνουν τα μέλη για την αντιμετώπιση ε, του νέου κύματο των μεταναστών. Εμεί ε, οι Ούγγροι πιστεύουμε ότι η Ουγγαρία θα πρέπει να αποφασίσει σαν χώρα τι πρέπει να κάνει για να καταπολεμήσει τα μεταναστευτικά προβλήματα διότι δεν έχουμε απεμπολίσει την κυριαρχία μας εμείς οι Ούγγροι σχετικά με αυτό. Είναι ένα καινοφανές φαινόμενο η μετανάστευση και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να νομοθετεί μόνο σε τομείς όπου ρητά έχει ανατεθεί την αρμοδιότητά της. Σύμφωνα με τις συνθήκες. Η μετανάστευση δεν είναι τέτοια πολιτική που εντάσσεται εκεί που θα πρέπει να τη χειρίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστούμε πολύ. Στη συνέχεια ο κύριος Τίμερμαν. Σας ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Τα καλύτερα μαντάτα σήμερα είναι ότι η κυρία Μόρβα απεκάλεσε αγαπητό τη ηγέτη τον πρόεδρο Γιούνκερ. Αυτό είναι κάτι το οποίο πράγματι για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να ε, ληφθεί υπόψη. Είναι όμως μια παρουσίαση, να το επεξηγήσω αυτό, του προγράμματος εργασίας Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τίποτα παραπάνω, τίποτα παρακάτω. Θα έχουμε επαρκή χρόνο στη συνέχεια να συζητήσουμε όλα τα στοιχεία του προγράμματος ε, εργασίας Ευρωπαϊκής Επιτροπής και δεν μπορώ σε σχέση με δηλώσεις για κάτι άλλο ή για μια μεγάλες ομολογίες που θα έπρεπε να γίνουν για θέματα πρέπει να εξετάσουμε επακριβώς εξειδικευμένα τις συγκεκριμένες προτάσεις που υποβάλλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να καταλήξουμε σε κοινά συμπεράσματα επ' αυτών. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό ως διεργασία και πιστεύω ότι καμιά φορά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λαμβάνει υπόψη αυτό το κοινοβούλιο πιο ε, σοβαρά από ότι κάποια μέλη στα άκρα, ε, ακραία μέλη ίσως ε, του Ευρωκοινοβουλίου αν θέλετε. Θα πρέπει λοιπόν να συμφωνούμε με το Κοινοβούλιο σε Επιτροπή ώστε να ευθυγραμμιζόμαστε με τα δικά σας, τις δικές σας κατευθύνσεις να λαμβάνονται κοινέ αποφάσεις που είναι αυτά που χρειαζόμαστε, αυτές που χρειαζόμαστε. Διαβάζοντας την έκθεση, νομίζω του ιδρύματο Μπέρτερσμαν, του Ιδρύματος Μπέρτελσμαν με παράθεμα σήμερα στην Ευρώπη 26 εκατομμύρια παιδιά και νέοι απειλούνται από τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό Αυτά θα πρέπει να κατευθύνουν το έργο και τις εργασίες μας. Αυτά πρέπει να αντιμετωπίζουμε με συγκεκριμένες πρωτοβουλίες. Ξέρετε πόσο υψηλή είναι η ενεργεία μεταξύ των νέων στα κράτη-μέλη μας. Για αυτούς τους λόγους χρειαζόμαστε και πρέπει να ακολουθήσουμε διαθωτικές ε, μεταρρυθμίσεις. Γι' αυτό πρέπει να δημιουργηθούν ευκαιρίες στην ενιαία εσωτερική ψηφιακή αγορά, στην εσωτερική αγορά. Γι' αυτό πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι πολίτες δεν θα εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν την ελευθερία κυκλοφορία ως απειλή απειλή εναντίον τους αλλά ως μια μεγάλη ευκαιρία για να δημιουργηθούν ε, σταδιοδρομίες και ευκαιρίες. Γι' αυτό πρέπει να υποβάλουμε τέτοιες προτάσεις που θα οδηγήσουν σε καλύτερη κοινωνική προστασία των Ευρωπαίων πολιτών. Εφόσον αυτό φυσικά επιτρέπεται ε, από τη δράση τη ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτούς τους τομείς. Γι' αυτό βρισκόμαστε εδώ, για να ακούσουμε τις απόψεις σας, για να βελτιωθούμε και να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Αλλά στο τέλος να πω τούτο. Συζητάμε έντονα και σε βάθος με το δικό σας θεσμικό όργανο, την Ευρωβουλή και το Συμβούλιο από πλευρά σα ε, τη Ευρωβουλή εκπροσωπήστε στο Συμβούλιο από τον κύριο Γκίντε Φερχόφστατ και ελπίζω ότι μπορούμε να καταλήξουμε σε συμπεράσματα μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων που θα καταδεικνύουν ότι έχουμε κατανοήσει τα μηνύματα των πολιτών μα, ότι πρέπει να βελτιωθούμε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί με τον τρόπο που προετοιμάζουμε το νομοθετικό έργο να αποφεύγουμε σφάλματα να αποφεύγουμε αυτά τα οποία ανέφερε η κυρία Ιντφελτ ότι καμιά φορά δηλαδή υιοθετούνται αποφάσει γνωρίζοντα απόλυτα τα καλά ότι αυτές οι αποφάσεις είναι καλές και σωστές διότι εκπροσωπούν ένα συμβιβασμό αλλά δεν είναι όμως ε, θετικές διότι όταν εφαρμόζονται στα κράτη-μέλη τότε οι επιχειρήσεις υποφέρουν ε, και γι' αυτό υπάρχουν προσφυγές στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Αυτά πρέπει να λάβουμε υπόψη. Να υπάρχουν καταλεπτός ε, μελέτες επιπτώσεων προτού ληφθούν αποφάσεις ώστε να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της υπερβολικής γραφειοκρατίας του γραφειοκρατικού άκου που επιβάλλεται στις επιχειρήσεις. Έτσι πρέπει να δράσουμε φυσικά η δράση μας θα πρέπει έτσι να κατευθυνθεί. Και σε αυτή τη φάση αυτό το εγχείρημα πραγματικά αντιμετωπίζει υπαρξιακές ε, ε, προκλήσεις. Όλα συνέρχονται. Η οικονομική κρίση, η δημοσιονομική κρίση, η κρίση προσφύγων, οι διεθνείς απειλές, η κλιματική κρίση και προκλήσεις. Όλα αυτά συνενώνονται και απειλούν την ίδια τη ζωή και ύπαρξη των Ευρωπαίων. Και το ευρωπαϊκό εγχείρημα πρέπει να δώσει απαντήσεις ε, Αυτό λοιπόν το πρόγραμμα εργασιών τη Ευρωπαϊκή Επιτροπής είναι τμήμα τη ευρύτερη, μεγαλύτερη απάντηση που πρέπει να δώσουμε σε όλε αυτέ τι προκλήσει. Ε, δεν θα είμαστε αποτελεσματικοί αν δεν δρούσαμε με αυτόν τον τρόπο ε, ω θεσμικό όργανο μέσα στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Είμαστε πρόθυμοι να συνεργαστούμε με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να είναι αποτελεσματικό το έργο μα προ όφελο των Ευρωπαίων πολιτών. Ευχαριστώ. Σε ευχαριστούμε κύριε Τίμερμαν. Εδώ ολοκληρώθηκε η συζήτηση πολύ.